για το λαό, για τη σταθεροποίηση της περιοχής, κάτι το οποίο όλους θα ωφελήσει φυσικά και εμάς. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος, καταληκτικές της συζητήσεως. Τέλος της συζήτησης, ψηφοφορία αύριο. Il punto η κυρία Άστον πάλι, υπεύθυνη για εξωτερικές υποθέσεις και θέματα ασφάλειας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για AIDS, HIV, σχετικά με τη συνάντηση που θα γίνει στη Βιέννη από τις 18 μέχρι τις 23 Ιουλίου. Δίνω αμέσως το λόγο στη Βαρόνια Άστον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα το να πάρω μέρος σε αυτή τη συνάντηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βοήθεια για το AIDS. 11 μέρες απομένουν πριν από την 8η διάσκεψη που θα οργανωθεί στη Γενέβη, στην Βιέννη, συγγνώμη. Οι άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν, η κατάσταση χειροτερεύει και ιδιαίτερα στις χώρες όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτές οι περίπλοκες καταστάσεις οδηγούν στην αύξηση των θυμάτων από το HIV και το AIDS, ιδιαίτερα εκεί όπου μολύνονται πάρα πολλές γυναίκες και παιδιά. Αυτοί που ζουν με, με τον ιό, είναι οροθετικοί, φοβούνται να το δηλώσουν σε πολλές χώρες. Σε χώρες όπου η ομοφιλοφιλία, σαν παράδειγμα, καταδικάζεται, οι ασθενείς φοβούνται την φυλάκιση και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις και τη θανάτωση. Θα πρέπει να γίνονται όμως σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων όλων, ακόμα και των ασθενών. Και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά επίσης τα δικαιώματά τους για την βέλτιστη δυνατή ιατρική βοήθεια σε επίπεδο ε, και σωματικό και ψυχολογικό. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να υφίστανται ε, διακρίσεις λόγω της κατάστασής τους. Εμείς γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό της ασθένειας αυτής για τον αποκλεισμό τους από τη χορήγηση ε, δικαιώματος ασύλου. Πολλοί διώχνονται από την εργασία τους, από τα νοσοκομεία τα ίδια και από τα σχολεία. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ορισμένα συμπεράσματα το Νοέμβριο του 2009 και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης έτσι ώστε να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω των εξωτερικών μας προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ελευθερία διακίνησης αυτών οι οποίοι ζουν ε, με τον ιό του AIDS. έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος αυτών οι οποίοι είναι μόνιμοι ή προσωρινοί σε μια χώρα. Και γι' αυτό τροποποιούνται και οι κανονισμοί τελευταία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και αυτό θεωρείται κάτι το θετικό. Τους τελευταίους μήνες οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Βρυξέλλες και σε άλλες χώρες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την ποινικοποίηση της, του σεξουαλικού προσανατολισμού σε χώρες όπως η Ουγγάντα, η Γκάνα κτλ. Και επίσης για τις συνέπειες που προκαλεί αυτός ο προσανατολισμός σε χώρες όπως η Σενεγάλη. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ομοφιλοφίλων, ανδρών και γυναικών και όλων όσων υποφέρουν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Κολάρσκα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βαρόνη, κυρία Άστον, που παρευρίσκεται εδώ, παρόλο που πολλοί άλλοι αυτή τη στιγμή βλέπουν τον αγώνα ποδοσφαίρου. Ωστόσο η συζήτηση αυτή είναι σημαντική γιατί είναι ένα ιδιαίτερο σεπόδινο θέμα και παρόλο που τελευταία έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στην ε, αντιμετώπιση στην, στην, και στην ε, θεραπεία της ασθένειας έχουμε μόνο πέντε χρόνια όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για να εμποδίσουμε την εξάπλωση του ιού και τις νέες μολύνσεις. Ο αριθμός των μολυσμένων ατόμων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, για παράδειγμα μεταξύ γυναικών και νεαρών κοριτσιών. Γι' αυτό με το ψήφισμά μας δηλώνουμε ότι υποστηρίζουμε τριών τύπων δράσεις. Καταρχήν νομικές δράσεις, ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε τις ε, χώρες που προσβάλλονται ιδιαίτερα από τον ιό του AIDS, ούτως ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να χαράξουν σημαντικά προγράμματα δράσης. Επίσης, να θεσπίσουν νόμους κατά των διακρίσεων για να προστατεύσουν τους νοσούντες και τους φορείς. Και επίσης δίνουμε μία έμφαση στο θέμα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ενημέρωση ούτως ώστε να αλλάξουμε μια κατάσταση διακρίσεων σε μια μετάβαση προς κατανόηση και αποδοχή. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για τις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και για τον ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο. Επίσης, πέρα από τη χορήγηση φαρμάκων, δίνουμε έμφαση στη σημασία ε, πρόσβασης σε ορισμένες ε, θεραπείες για παράδειγμα στον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών με την Ινδία. Εδώ ανέκυψαν σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα το γεγονός ότι η Ινδία ε, παρασκευάζει ε, σκευάσματα χαμηλού κόστος για την αντιρετρογική θεραπεία και αυτή τη στιγμή ίσω υπογραφεί συμφωνία θα περιοριστεί η παραγωγή αυτών των σκευασμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κάσμαν έχει το λόγο για τρία λεπτά εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Βαρόνη, ακούγοντα τα εισαγωγικά τη λόγια, μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ότι μπορώ να πάω σπίτι μου, γιατί η δουλειά μου έχει γίνει. Σπάνια έχω ακούσει κάποιον ε, σε αυτή την πλευρά να ε, κατανοεί όχι μόνο αυτό το οποίο κάναμε, αλλά και αυτό το οποίο, όχι μόνο αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε να προστατεύσουμε εκείνου που είναι ιδιαίτερω ευάλωτοι. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να λάβει μια σωστή ε, προσέγγιση γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ενισχυθούν και να προστατευθούν και από τη δική της πλευρά και από την κυβέρνηση. Και Αναφέρουμε επίσης την αναθόρηση των στόχων της χιλιετίας. Δυστυχώς με τον ιό του AIDS ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Πάνω από 33 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν με τον ιό του AIDS. Το 2008 μόνο 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς στην υποσαχάρια Αφρική και οι περισσότεροι από αυτούς, το 60% είναι γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Έτσι λοιπόν είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα άτομα ως προς τις ίδιες επιλογές, ε, τις ίδιες επιλογές ως προς την χρήση του σώματός τους. Ε, θα πρέπει ε, να ενισχύσουμε επίσης τους ομοφιλόφιλους ή τους τρανσέξουαλ, οι οποίοι ε, δεν έχουν συχνά αυτή την επιλογή. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερόμεθα ε, προς εκείνους που προσβάλλονται από όλες αυτές τις διακρίσεις. Υπάρχουν υψηλά επίπεδα μόλυνσης μεταξύ των όσων, ε, μεταξύ των ομοφιλοφίλων που αρνούνται την ίδια τους τη σεξουαλίτη λόγω της χαμηλής τους αυτοπεποίθησης, επίσης μεταξύ των χρηστών, μεταξύ των προσφύγων και μεταξύ των μετακινούμενων εργαζόμενων και όσους παρέχουν ε, σεξ ε, ε, ως επάγγελμα. σε πολλές χώρες η νόση προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Αλλά δεν είναι μόνο αρνητική αυτή η ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τη προσοχή σε αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι πίσω από αυτά τα στατιστικά στοιχεία των εκατομμυρίων ε, ε, κρύβονται αληθινές ζωές ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από το AIDS, που έχουν χάσει τη ζωή τους, που έχουν χάσει την οικογένειά τους, ε, τα αδέλφια τους κλπ. Ζωές που καταστρέφονται λόγω της απώλειας των οικείων τους υπάρχει μια πλήρης ε, απώλεια και σπατάλη της ανθρώπινης ζωής λόγω της ε, προβλέψιμης εξάπλωσης του ιού του AIDS. Μια εξάπλωση την οποία όμως δεν κάναμε αρκετά για να την αποφύγουμε. Ευχαριστώ Δημοκρατική και Φιλελεύθερο κύριο Συμβέλτη για τέσσερα λεπτά. Κύριε Βέλτε, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη Βαρόνια Άστον για την εισαγωγή που έκανα αλλά και τους, ε, συναδέλφου συναδέλφους μου για τα λόγια που πρόφεραν. Θα ήθελα να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα τα όσα υπόθηκαν πριν από λίγο. Ο Μάικ Κάσουιν είπε ότι είναι μια προβλέψιμη, μια δυνάμενη να προληφθεί νόσος με πολύ απλά μέσα, δωρεάν, δεν κοστίζει δεκάρα. Θα μπορούσαμε να προλάβουμε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις ε, AIDS. Θα μπορούσαμε να προλάβουμε τόση δυστυχία. Ας δούμε μερικές λέξεις κλειδί. Το στίγμα. Ο κύριο, η κυρία Κολάσκα αναφέρθηκε στο θέμα των ε, διακρίσεων. Αναφερθήκατε και εσείς αυτό, κυρία Άστον. Ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το στίγμα. Σκεφτείτε ότι ότι σε αρκετές χώρες μέλη δεν επιτρέπεται στους ομοφιλόφιλους να είναι αιμοδότες. Υπάρχουν χώρες μέλη που ενάντια σε όλους τους νόμους, ενάντια σε όλες τις αρχές ζητούν σε κάποιον να, να κάνει ε, μια δήλωση ότι δεν έχει έτσι πριν να μπει στη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από το στίγμα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το ιστενοκεφαλιά όταν τίθεται το θέμα της σεξουαλικής ηθικής αν θέλετε. Με σοκάρει όταν διαπιστώ τόνο, ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα που θεωρούν ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ψήφισμα γιατί γίνεται αναφορά στα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Απλά και μόνο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις αρχές, αυτές τις έννοιες. Αν είχαμε τη στήριξη όλων των μελών θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε τόση μα τόση δυστυχία και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να, να αρνηθούν προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να μπορούν να κοιτάνε ανθρώπους στα μάτια και κυρίως γυναίκες που πάσχουν από ένα τέτοιο νόσημα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να τονιστεί. Η θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνε για το σώμα τους. Οι γυναίκες είναι εκείνες που αποφασίζουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι πράγματα που δεν κοστίζουν δεκάρα. Δεκάρα δεν κοστίζουν. Πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και σε φάρμακα. Μιλάμε για βασικά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Περί αυτού πρόκειται. Ε, και όμως αυτό το δικαίωμα το αρνούμεθα σε ορισμένους ανθρώπους. Ή τους το δίνουμε λες και πρόκειται για χάρη, λες και πρόκειται για προνόμιο. Είμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που πλήττει χώρες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα Μία, ένα υγιές εργατικό δυναμικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη. σε επενδύσουμε στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω έκκληση στις χώρες αυτές ε, που προβλέπουν περικοπές στον προϋπολογισμό στον ε, τομέα αυτό, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. <coughs> θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Δεν πρέπει να μιλάμε για περικοπές θα πρέπει βεβαίω να αναλάβουν, και την ευθύνη του οι εθνικές κυβερνήσεις. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα μέλη όλων των ομάδων να υποστηρίξουν αύριο το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε ονόματο των Πρασίνων Αουτάλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Υποστηρίζω αγκαρδίως αυτά που είπαν οι τρεις συνάδελφοι από τις άλλες πολιτικές ομάδες για το HIV και το AIDS. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Άστον. Το ψήφισμα το οποίο θα υιοθετήσουμε αύριο θα είναι μια σημαντική συνεισφορά στη 18η διάσκεψη η οποία θα οργανωθεί στη Βιέννη στο τέλος του μήνα. Εκεί θα μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες ακολουθούν ακόμα πολιτικές που στοιχειοθετούν εμπόδια σε αυτούς και στη ζωή αυτών που υποφέρουν από AIDS. Και λειτουργούν επίσης και σαν εμπόδια, σαν εμπόδια στην πρόληψη αυτής της ασθένειας. Λέμε εμείς ότι υπάρχουν 106 τέτοιες χώρες στον κόσμο. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα και βασικό στόχος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Να υπογραμμίσουμε δηλαδή ότι απαιτούνται πολιτικές καταπολέμησης του HIV και του AIDS συγκροτημένες, να τεθεί τέρμα στις διακρίσεις και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να ποινικοποιούν την ομοφιλική συμπεριφορά. Θα πρέπει να πούμε στις χώρες αυτές ότι αυτό δεν θα πρέπει να, να λαμβάνονται αποφάσεις επί τη βάση των παραδόσεων μόνο, αλλά θα πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών των χωρών τους. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Αριστερά, Ματίας, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Άστον, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν μέχρι τώρα. Εκατομμύρια νεκροί υπήρξαν το 2007, εκατομμύρια και τώρα και οι αριθμοί αυτοί δυστυχώς αυξάνονται και υπάρχουν και εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων που υποσφέρουν από το HIV και δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ε, σε ιατρική φροντίδα. Στην υποσαχαρική Αφρική είναι επίσης εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι αποφέρουν. Ο αριθμός των γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Και θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο την πρόληψη κυρίως και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. θα πρέπει το θέμα αυτό να καταστεί προτεραιότητα στην προστασία της δημόσιας υγείας και να καταπολεμηθούν όλες οι διακρίσεις που υφίστανται οι ασθενείς και στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν παράδειγμα, εμοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν το ευεργετικό τους αυτό λειτουργήμα επειδή έχουν συγκεκριμένους σεξουαλικούς προσανατολισμούς. θα πρέπει να αυξηθούν οι πιστώσεις για την καταπολέμηση της ασθένειας και η μείωσή τους θα χειροτερεύσει την κατάσταση. Στην Ευρώπη λέμε ότι είμαστε πρότυπο για τη βοήθεια για την ανάπτυξη και δεν πρέπει να είναι απούσα η Ευρώπη από αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους υπολείπους εγγεγραμμένους. Ο κύριος Κέλλη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Βαρόνη Άστον για την εξαιρετική της δουλειά και για τις απαντήσεις που έδωσε με πολύ σωστό τρόπο στη σύντομη παρουσία της εδώ σήμερα. Ασχολούμαι με το θέμα εδώ και λίγα χρόνια όταν είχα πάει εθελοντικά στο Μαλάουι. Είδα την καταστροφή που έχει προκαλέσει η ασθένεια αυτή εκεί, στα παιδιά και στους ενήλικες. Είναι μια χώρα 12 εκατομμυρίων προσδόκιμο ζωής είναι 32 χρόνια μόνο. Και το υψηλότερο ποσοστό ασθενών από HIV και AIDS. 25% των παιδιών είναι άρρωστα. 60.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο και 80.000 ασθενούν από HIV. Και δυστυχώς μόνο το 30% έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο, στην τριπλή θεραπεία. Τι απαιτείται λοιπόν πρώτον ιατρική βοήθεια, δεύτερον πρόληψη και τρίτον η θεραπεία όταν, και τρίτον μάλλον η εκπαίδευση έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόληψη και θα πρέπει να έχουμε και μια πιο ανθρώπινη στάση απέναντι στους ασθενούς. Η κυρία Στον αναφέρθηκε στο θέμα της απομάκρυνσης ορισμένων πρακτικών που λόγω ακριβώς ε, της, ε, των πρακτικών που ακολουθούν ορισμένες φυλές δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα στις γυναίκες και στα παιδιά και κάποιες τέτοιες παραδοσιακές πρακτικές θα πρέπει να καταδικαστούν. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις αρχές των χωρών γιατί αυτό που παρατήρησα στο Μαλάουι διαβάζοντας την εφημερίδα διάβασα πολλά άρθρα που ασκούσαν κριτική στις ΜΚΟ γιατί δεν είχαν καταφέρει να συνεργαστούν με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απαιτείται λοιπόν να απομακρύνουμε τον απικιακό, τον απικιακό θα έλεγα πατερναλισμό και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς να απαλλαγούν από τη μάστιχα του HIV. Λούνατσεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε ένα κοινό ψήφισμα. Ελπίζω με την πλειοψηφία του σώματος να ψηφιστεί. Γιατί ελέγχθη για την προετοιμασία της 18ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης στη Βιέννη, που είναι η, χώρα, η πόλη όπου ζω, ε, είναι, το θέμα είναι εδώ και τώρα Κάτι το οποίο δεν κάναμε στο παρελθόν, γιατί όπως ελέγχθη από όλους τους ομιλητές εδώ, το HIV και το AIDS οδηγεί στο αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που είναι φορείς, έχουν μολυνθεί από τον ιό ή νοσούν, θεωρούνται ως περιθωριοποιημένα άτομα, όχι σαν κάποιοι που είναι κανονικά ενταγμένοι στην κοινωνία. Και συνεπώς υπάρχει η ανάγκη να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτούς τους ανθρώπους, την πρόληψη και την ε, παροχή ε, φροντίδων υγείας. Εάν ο ΠΟΕ στην δήλωση της Ντόχα το 2001 δήλωσε σαφώς ότι η υγεία προηγείται των εμπορικών συμφερόντων, κάτι που είναι ιδιαίτερο σημαντικό στην Αφρική, όπου 60% των μολυσμένων ατόμων είναι γυναίκες, άνθρωποι που κατά παράδοση έχουν μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και έχουν λιγότερα χρήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν τα φάρμακα για το AIDS να είναι προσβάσιμα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, οι γυναίκες και τα νερά κορίτσια ε, μολύνονται πολύ περισσότερο από την έναρξη της επιδημίας, ε, της νόσου. Ε, ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από όλου και ήθελα να κάνω έκκληση και προ εκείνους που μέχρι στιγμής δεν προσυπέγραψαν το, τη δήλωση να υπερψηφίσουν το ψήφισμα ούτω ώστε τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και σεξουαλικά δικαιώματα να κατοχυρωθούν για όλους ιδιαίτερα ε, για όσους έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS. Ευχαριστώ. Το λόγο στον κύριο Νίκολα Σέικ. Δύο λεπτά. Παρόλε τι ιατρικέ γνώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, το πρόβλημα με το AIDS ε, εμένει. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι περισσότεροι προσβάλλονται από την νόσο αυτή σαν αποτέλεσμα του ότι κάνουν σε χωρίς προφυλάξεις. Πώς διαδίδεται, πώς μεταδίδεται αυτή η νόσος. Άτομα που έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις ή ε, άτομα που παρέχουν πληρωμένο έρωτα. Ας μην είμαστε όμως αφελείς. Ας μην υποκρινόμαστε ότι ο ιατρικός έλεγχος μία φορά την εβδομάδα θα λύσει το πρόβλημα. Είμαι γιατρός ο ίδιος και ξέρω ότι ακόμα κι αν επισκέπτεται κάποιος ένα γιατρό μία φορά την εβδομάδα το πρόβλημα δεν λύνεται. Όπως είπαμε, μία ευάλωτη ομάδα είναι οι ομοφιλόφιλοι, όπως γνωρίζουμε στην κοινότητα των ομοφιλοφιλών το ποσοστό του ε, AIDS είναι πάρα πολύ υψηλό. Επίσης, το να έχει κανείς πολλούς ερωτικούς τριντρόφους. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνουν έρευνες σε νέα Α, φάρμακα. Τα αντιϊκά φάρμακα δεν είναι πλέον αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Ελπίζουμε να βρούμε νέα μόρια που θα μας επιτρέψουν να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ είμαι υπέρ του να βοηθήσουμε την Αφρική με κάθε δυνατό τρόπο. Εκεί υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν προσβλήθει και θα πρέπει ιδιαίτερα στην υπος ε, Σαχάρη Αφρική να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η δικασία άλλη, κύριος Σαλβατόρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ το AIDS αποτελεί απειλή για την υγεία όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών. Κάθε χρόνο πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι και το πρόβλημα αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στις αναπτυσσόμενες κοινότητες. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε. Χρειάζεται ακόμα περισσότερη πρόληψη, ακόμα περισσότερη ενημέρωση αλλά κυρίως χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις οικογένειες γιατί το πρόβλημα του νοσούντος από έτσι είναι πρόβλημα μιας ολόκληρης οικογένειας. Θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να υιοθετήσουν έναν πιο ε, σωστό τρόπο ζωής. Στόχος είναι η προβληματική και αυτή, ε, το πρόβλημα αυτό να μειώνεται όλο και περισσότερο όσο περνάει ο χρόνο. Κύριε είναι ιδιαίτερος ε, οι νέοι άνθρωποι που υποτιμούν τον ε, κίνδυνο της νόσου. Ε, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερβολικά νέοι για να ε, θυμούνται την ενημερωτική εκστρατεία της δεκαετίας του 80 και το AIDS, οι κίνδυνοι του AIDS δεν διδάσκονται στα σχολεία. Σε μία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου είχαμε σαν αποτέλεσμα ότι οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν μία ισχυρότερη ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νόσου. Ε, θα πρέπει επίσης να ε, καταπολεμηθούν, ε, κατακολουθεί η άχνοια στον πληθυσμό και οι αναλυθείς πληροφορίες. θα, πρέπει, θα πρέπει να, επίσης να παρεμποδίσουμε ένα στιγματισμό των νέων ατόμων που μολύνονται από την όσο. Τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το είπε και η κυρία Γουέφμαν προηγουμένως. Παρότι 33 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι παγκοσμίω είναι σήμερα φορείς του θανατηφόρου ιού, πολλοί είναι εκείνοι ιδίω οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ε, τους κινδύνους που ε, συνεπάγεται ε, η έλλειψη προσοχής και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να συνεχίσουμε τις εκστρατείες ενημέρωσης και πράγματι η ένταση που υπήρχε στο παρελθόν δεν υπάρχει σήμερα. ένα δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που εγκυμονεί γνωστοποίηση της μόλυνσης και που έχει ως αποτέλεσμα περίπου το 30% των ατόμων στην ευρωπαϊκή ένωση που πάσχουν να μην γνωρίζουν ότι είναι φορείς με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης. με γνώμονα αυτούς τους δύο στόχους πρέπει ο ιός να αντιμετωπιστεί ως παγκόσμια προτεραιότητα υγεία η επιτροπή και το συμβούλιο να δράσουν υπεύθυνα και να προωθήσουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων είναι καθοριστικό αυτό να δοθεί έμφαση στην καθοδήγηση και ενημέρωση των νέων και τέλος το κοινό να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί σωστά προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο κοινωνικός αποκλεισμό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η διάσκεψη της Βιέννης θα ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών να προστατευθούν από τις συνέπειες της μόλυνσης αυτής και θα πρέπει να τύχουν ε, εξαιρετικού επίπεδου ε, στο μέλλον ιατρικής βοήθειας. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα διατηρήσουμε την προσπάθειά μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και στο εσωτερικό της Ευρώπης και σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες και κοντά στα σύνορά μας και σε ε, μακρινές ε, υπήρους. Θα είμαι στη Μέση Ανατολή και δεν θα μπορέσω να είμαι στη διάσκεψη της Βιέννης, αλλά ο Επίτροπος Ντάλι που είναι υπεύθυνο για τα θέματα υγείας θα αντιπροσωπεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πάρει μέρος στην εναρκτήρια συνεδρίαση και θα ομιλήσει. Πολλές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από διάφορους τομείς της ανάπτυξης, της υγείας κτλ. θα πάρει μέρος επίσης. Και οι οδήποτε μέλος συμμετέχει σε αυτή τη διάσκεψη τους καλώ να συναντήσουν τις υπηρεσίες μας στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα οργανωθούν και δορυφορικές συνεδριάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνοντας θα ήθελα να πω κάτι το οποίο έχετε κάνει και εσείς. Σήμερα έγινε ένας ε, σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας στην Νότια Αφρική και θυμήθηκα την Νότια Αφρική που είχα πάει πριν λίγα χρόνια. Ε, με οδηγούσαν με αυτοκίνητο έξω από τον Τζοχάνεσμπεργκ και αυτός που οδηγούσε μου συζητούσε για τα προβλήματα του HIV και του AIDS στη χώρα αυτή. Ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν πολλοί, μεταξύ των οποίων και μία τραγουδίστρια πολύ γνωστή, η Άννη Λένοξ. Και περάσαμε, μου είπε διάλεξε ένα χωριό για να δεις τι ακριβώς γίνεται και έδειξα ένα χωριό και μπήκαμε μέσα στο χωριό και με οδήγησε στο νεκροταφείο. Και είπε, ξέρεις, στην Αφρική η παράδοση είναι να μην βάλει κανείς ταφόπλακα ε, ε, τα φόπλακα αν δεν περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή της ταφής, την μέρα της ταφής. Και πήγα λοιπόν σε αυτό το νεκροταφείο και τι είδα. Εκατοντάδες τάφους χωρίς ε, πλάκες και μου είπε ότι όλοι αυτοί ουσιαστικά πέθαναν από AIDS. Μιλάμε για μια καθόλου απαραίτητη καταστροφή και ελπίζω ότι θα μπορέσω να κάνω και εγώ ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Άστον, κλείνει η συζήτηση αυτή. Περνάμε τώρα στην δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπα του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, γιατί